στην ΕΡ μια νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισηγήτρια έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε. Τα δάση μας και η δασική βιομηχανία ε, συμβάλλουν στην απασχόληση αλλά εξασφαλίζουν βιωσιμότητα, ποιότητα ζωής ε, και δημιουργία αξίας με 3,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας είναι στην τρίτη θέση στην απασχόληση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μετά τους κλάδους της μεταλλουργίας και των τροφίμων. Περισσότερες από 400.000 επιχειρήσεις που στηρίζονται στη δασοκομεία συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη σε ποσοστό 7% ενώ εκμεταλλεύονται μόνο το 60% της ε, ετήσιας δασικής ανάπτυξης. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό σπόρο η ξυλία με μεγάλη οικονομική σημασία για τι αγροτικέ περιοχέ και όχι μόνο. Με την προσεκτική μέρημνα και διαχείριση των ευρωπαϊκών δασών ε, και των άνω των 16 εκατομμυρίων διοκτητών δασών διασφαλίζεται ότι τα δάση είναι σε θέση να εκπληρώσουν τι οικολογικέ, οικονομικέ και κοινωνικέ λειτουργίε του με βιώσιμο τρόπο. Άνω των 50% των ευρωπαϊκών δασών είναι ιδιοκτικέ ιδιοκτησίε. Ο στόχος λοιπόν είναι η δασική πολιτική ε, να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε το θέμα των ε, πόρων στην Ευρώπη. Ε, το βασικό στοιχείο, ένα βασικό στοιχείο στην έκθεση είναι ο καλύτερος συντονισμός. Η ενέργεια, το περιβάλλον, το κλίμα ε, επηρεάζουν πολύ τη διαχείριση των δασών που θα πρέπει στις διάφορες ευρωπαϊκές στρατηγικές να έχουν καλύτερη θέση λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα των κρατών μελών. Νέες σε γραφειοκρατικές εφαρμογές στη δασική πολιτική δεν θα ε, γίνουν δεκτές. Το Κοινοβούλιο τάσεται υπέρ του διαχωρισμού των ε, σχεδίων για τα δάση στο Natura 2000. Ε, δεν ε, θα πρέπει να ε, υπάρξει μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την κατάρτιση, κατάρτιση σχεδίων στο πλαίσιο της Natura 2000 στους ιδιοκτήτες δασών. χρειάζεται να υπάρξουν κριτήρια βιωσιμότητας. Επίση, σημαντικά είναι τα κριτήρια τα οποία θα ισοδυναμούν με ποιοτικά κριτήρια και θα πρέπει πάντα να ισχύουν για το σύνολο του τομέα. Είναι ε, σημαντικό να μην υπάρχει μια σειρά κριτηρίων που θα εφαρμόζονται παντού, ε, αλλά να υπάρχουν ε, τα κριτήρια του Forest Europe ως βάση για μια στρατηγική βιωσιμότητας. Επίσης, ε, ιδιαίτερη προσοχή ε, θα πρέπει να δοθεί στους λεγόμενους κατάντι κλάδους της βιομηχανίας που μπορούν να επωφεληθούν από αποδοτικές δυνατότητες και ε, σημαντικό είναι να έχουμε έμφαση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση. Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι επίσης πολύ σημαντικά και έχουν τονιστεί πολύ νέες δυνατότητες παραγωγής ε, είναι ο στόχος μας για να υπάρξει εξέλιξη στη βιοοικονομία, ε, αλλαγή του βιώσιμη αξιοποίηση των πρώτων υλών ε, για να έχουμε συμβολή στο καλύτερο περιβάλλον και το κλίμα πιστεύω ότι χρειάζονται επενδύσεις, η μόνιμη δασική επιτροπή πρέπει να ενισχυθεί, ε, η εντολή της να αναβαθμιστεί και να συμμετέχουν περισσότερο τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους στην Επιτροπή Γεωργίας συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά, ε, ιδιαίτερα και η γνωμοδότηση από την Επιτροπή Βιομηχανίας και Περιβάλλοντος ενίσχυσαν ε, την έκθεση και ε, στήριξαν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βοηθοί επίσης συνεργάστηκαν με τρόπο πολύτιμο όπως και οι γραμματική ο γραμματέας τη Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ για τη συνεργασία όλων. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο Κέστιγκερ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Και εδώ ζήτησαν πάρα πολύ το λόγο, υπερβολικά μεγάλος αριθμό. Θα δώσω το λόγο μόνο ε, στους συναδέλφους που δεν έλαβαν το λόγο νωρίτερα. Η κυρία Νόιχελ πρώτη. Ευχαριστώ πολύ να πω δύο λόγια για τη νέα δασική στρατηγική είναι σωστό και σημαντικό η δασική πολιτική, ιδίω σε εθνικό επίπεδο. Σημαντικό και αναγκαίο είναι όμω ιδιαίτερα όταν οι προκλήσει είναι διασυνοριακέ για τα δάση να σκεφτόμαστε και να τα δρούμε ευρωπαϊκά. Πολλά είναι σε καλό δρόμο και στηρίζω την συνάδελφο Κέστιγκερ σε πολλά θέματα. Ε, θα πρέπει να δούμε τα οικονομικά, κοινωνικά θέματα και τα περιβαλλοντικά θέματα και θα πρέπει βεβαίως να ε, ταχθούμε υπέρ της βιωσιμής ανάπτυξης. Όλα αυτά προχωρούν καλά, αλλά έχουν μείνει ανοιχτά θέματα. Τρία θα αναφέρω. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν κριτήρια ευρωπαϊκά για τη βιωσιμότητα. Απαραίτητο είναι να προβληματιστούμε για το δάσος το οποίο αυξάνεται αλλά υπάρχουν, ε, υπάρχει ανάγκη για ε, καλύτερη διατύπωση της χρήσης που θα γίνει στο δάσος. Όχι και ε, με την ε, επίπτωση που θα έχει κάθε χρήση. Χρειάζεται καλός συντονισμός και αυτόν θα ήθελα να ζητήσω για το άμεσο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ κυρία Νόχελ και τώρα ο κυρίος Τσαμπάτσκι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ παρά να εγκρίνω η νέα δασοκομική ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια προσέγγιση συστηματοποιημένη. Νομίζω ότι η δασική πολιτική πρέπει να είναι μια εθνική προτεραιότητα και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν κοινοτικέ ρυθμίσεις. Ωστόσο, ορισμένα κοινά μέτρα είναι απαραίτητα και επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί προστιθέμενη ε, ε, αξία. Στη χώρα μου έχει προβλήματα ο τομέας. Τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά χρησιμοποιούνται για παράνομες χρήσεις ε, και η παραγωγή, η παράνομη ξυλίας εξάγεται σε τρίτες χώρες. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια ενώπιον αυτών των παρατυπιών και παρανομιών. Θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις, ώστε ο τομέας να μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερη προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ κύριε Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά την κυρία Κέρστινγκερ για αυτή την έκθεση πρωτοβουλία με τις 28 τροπολογίες. Είναι ισχυρό το πολιτικό μήνυμα για τους ιδιοκτήτες δασών και τη δασική οικονομία. Είναι σημαντικό τα δικαιώματα ιδιοκτητών των 16 εκατομμυρίων ιδιοκτητών δασών να ενισχυθούν και να διατηρηθούν, να διασφαλιστούν. Δεν επιτρέπεται να ε, ε, αναλάβουν αρμοδιότητες ε, για την κατάρτιση σχεδίων και συμφωνούμε με τη... και, δεν συμφωνούμε με το να αναλάβουν αρμοδιότητες στα πλαίσια του Νοτρό 2000. Η, δασική πολιτική είναι σημαντική για την εργασία, την απασχόληση και προφανώς ε, συμβάλλει στην διατήρηση του κλίματος. Ε, καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει την έκθεση αυτή πρωτοβουλίας στην ε, δασική της στρατηγική. Ευχαριστώ κυρία Μούλερ. Και τώρα η συνάδελφος Κούμπουλα Νάτρη. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι το γεγονός ότι ε, τόσο αργά μέσα στη μέρα ασχολούμεθα με αυτό το θέμα δεν σημαίνει ότι ε, δεν ενδιαφερόμεθα για αυτό το θέμα. Στη Φιλανδία είναι τεράστια οι δασικοί, τεράστιες οι δασικές εκτάσεις που πρέπει να προστατευτούν όπως το Βέλγιο. Ε, πρέπει να προστατεύσουμε τους φυσικούς μας πόρους ε, να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη ε, για τα καύσιμα, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική ε, αλλαγή. Η οικονομία, ε, δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα, πρόγραμμα, ένα σχέδιο δράσης. Ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν μια συνεκτική προσέγγιση για να δούμε όλες τις δυνατότητες και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τη βιοοικονομία και να κάνουμε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε ώστε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη τεχνογνωσία στην ε, επεξεργασία και να διατηρήσουμε και τα πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που έχουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η συνάλφος Μακιντάιρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Κούστιγκερ για την έκθεσή της. Νομίζω ότι η βιώσιμη διαχείριση περιορίζεται από νομοθεσία γραφειοκρατική, υπερβολική όπως η ρύθμιση για την ξυλία. Γι' αυτό χαίρομαι ότι διότι προτείνει η έκθεση αναθεώρηση της νομοθεσίας για την θέσπιση μιας νέας νομοθεσίας με λιγότερες απαιτήσει. Καταλαβαίνω την ανάγκη να εφαρμόζεται η ρύθμιση εισαγωγές τρίτων χωρών, αλλά μια γενική δεν είναι απαραίτητη. Χρειάζονται στοχοποιημένες πρωτοβουλίες και διαδικασίες ούτω ώστε ε, η ξυλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιβαρύνεται με υπερβολικό κόστος και υπερβολική γραφειοκρατία. Ευχαριστώ και τέλος ο συνάλθος Μπράνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να μιλήσω για την σημασία της δασοκομείας των δέντρων και της ξυλίας για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα βλέπει κανείς τις αλλαγές δημιουργεί θέσεις εργασίας και βελτιώνει την υγεία. Σχετικά με την κλιματική αλλαγή απορροφούμε 10% των εκπομπών σε, σε, λόγω έλλειψης δασικής κάλυψης. Αν μπορούμε να αυξήσουμε την κάλυψη στην Ιρλανδία θα περάσουμε από 10% σε 18% μέχρι το 2050. Έτσι θα μπορέσουμε να δεσμεύσουμε περισσότερο άνθρακα και να μειώσουμε την κλιματική αλλαγή. Επίσης νέες θέσεις εργασίας στον τομέα στην δική μου μου ε, περιοχή βορειοανατολικά υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και μπορούν πάρα πολύ να εργαστούν στον δασικό τομέα και η βελτίωση της υγείας για τους τρεις αυτούς λόγους βλέπουμε ότι ο καλύτερος φίλος ε, του ανθρώπου δεν είναι ο σκύλος αλλά είναι το δέντρο. Ευχαριστώ συνάδελφε Μπράνεν. Ολοκληρώνεται η συζήτηση με την ε, παρέμβαση του Επιτρόπου Χόγκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Παρά το γεγονός ότι είναι περασμένη ώρα, χαίρομαι που συζητούμε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα και χαίρομαι που εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδέλφους που συμμετέχουν στη διαδικασία για την εφαρμογή της νέας πολιτικής για τα δάση κυρίως ο Επίτροπος Βέλα, ο ε, Επίτροπος Κανιέτε, ε, για να αναφέρω κάποιους εξ αυτών. Ε, τρόπον όλοι ενδιαφερόμαστε για το θέμα το αυτό, γι' αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως την εισηγήτρια, την κυρία Κρέσιγκερ, για την τόσο σημαντική έκθεση και φυσικά και τους και εισηγητές. Χαιρόμαστε που συζητήθηκε και στην Επιτροπή ΕΜΒΗ και στην Επιτροπή ΕΤΡΕ μια τόσο σημαντική έκθεση. Το γεγονό ότι δεν υπάρχει κοινή δασική πολιτική στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε μακρά ιστορία συνεισφοράς στην εφαρμογή των πολιτικών των κρατών μελών για τα δάση βάσει τη αρχής της επικουρικότητας. Έχουμε κοινούς στόχους και κοινέ αξίες για την εφαρμογή της δασικής πολιτικής. Η δασοκάλυψη είναι πολύ μεγάλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένω είναι πάρα πολύ σημαντική για την οικονομία και για την κοινωνία μα. Πολλές ε, ε, πτυχές βοηθούν στη δασική πολιτική, η ανάπτυξη της υπαίθρου, ε, η βιοενέργεια, η βιοοικονομία και μέσω αυτών των πολιτικών η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια πολύ σημαντική συνεισφορά για την εφαρμογή της βιώσιμης δασικής διαχείρισης και αποφάσεις των κρατών μελών που σχετίζονται με τα δάση και το συνολικό δασικό τομέα, καθώς επίσης και την προστασία των δασών. Και από πολιτική σκοπιά θα ήθελα να επισημάνω ότι η νέα στρατηγική για τα δάση ε, είναι, ε, έχει σύμπνοια με την ε, πολιτική της Επιτροπής Γιούγκερ και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο δασικός τομέας εκπροσωπεί το 7% του μεταπητικού τομέα ΑΕΠ και κυρίως το γεγονός ότι σε απομακρυσμένες περιοχές δημιουργεί θέσεις εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μια χώρα όπως η Φιλανδία, να επενθυμίσω ότι όταν ε, συμπεριλάβαμε τον χαρτοπολτό και στο, το χαρτί, ε, αυξήθηκαν οι εξαγωγές στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά τα περιβαλλοντικά ωφέλη ε, είναι πολύ σημαντικά για όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο για το κράτος μέλος που ε, εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε σωστή διαχείριση για τους φυσικούς μας πόρους και θα συνεχίσουμε να έχουμε αποτελέσματα και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή. Η στρατηγική βασίζεται και στην κλιματική αλλαγή ως ένα τρόπο να μετριάσουμε τις συνέπειες του περιβάλλοντος, τη βιοπικιλότητα, ε, διότι διαδραματίζει και αυτή πολύ σημαντικό ρόλο για την ε, βιοπικιλότητα ε, και μας ενδιαφέρουν οι δασικές περιοχές. Η βιομάζα είναι πάρα πολύ σημαντική, επομένως και στην ενέργεια έχουμε συνεισφορά από τα δάση. Αλλά υπάρχουν και άλλοι ευρύτεροι τομείς, ε, τομείς καινοτομία, ανάπτυξη δεξιοτήτων που βοηθούν σε μια βιώσιμη βιοοικονομία. Όπως σας είπα, τα δάση διαφέρουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Φιλανδία στη Μάλτα, από την Πορτογαλία στη Ρουμανία. Επομένως, η αρχή της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της καλύτερης νομοθεσίας θα βρίσκονται στο επίκεντρο της εφαρμογής της ε, στρατηγικής για τα δάση. Αν εξετάσουμε την ίδια τη στρατηγική, ο στόχος είναι να καθορίσει ένα πλαίσιο για δράσεις που βασίζονται στα δάση με βάση το συντονισμό των διαφόρων πολιτικών ε, των κρατών μελών για τα δάση και να υπάρχουν και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με δραστηριότητες για τα δάση. Η στρατηγική παρέχει μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση των δασών και επικεντρώνεται στα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη των δασών συνδυάζει εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα δασικής πολιτικής και αξιολογεί όλη την αλυσίδα της δασικής πολιτικής, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και συνεισφορά σε θέσεις εργασίας και κυρίως σε περιοχές της υπαίθρου. Ε, με βάση λοιπόν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Στρατηγική για τα Δάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και του ενδιαφερομένου αναπτύσσει ένα πολιετέ στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τι συγκεκριμένε δράσει που θα πρέπει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, αλλά κυρίω να διαπιστώσει ποιο είναι το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή. Γι' αυτό ακριβώ και θα έχουμε και συμμετοχή των ε, ενδιαφερομένων μερών θα υπάρξει συντονισμός των διαφορών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και τη διαδικασία ε, εξέτασης και απολογισμού της κατάστασης. Ε, θα λάβουμε υπόψη μας βεβαίως και την έκθεσή σας ε, στην προετοιμασία του πολιετούς διαχειριστικού προγράμματος για τη στρατηγική για το ΓΑΣ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η